Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να ζητήσω από τους συναδέλφους να καλωσορίσουν από το Εύρο Μαϊντάν μια αντιπροσωπεία που έφτασε σήμερα το πρωί. Έφυγαν από το Κίεβο χθε το βράδυ και θα χαρούν να συναντήσουν όσο περισσότερους μπορούν από εσάς. Ε, είναι ε, πάνω ε, πίσω μου. Είναι οι άνθρωποι που δίνουν ειρηνικές, όχι βίαιες μάχες στους δρόμους του Κιέβου. on this? No. no, Yeah, because it's. Uh... We did a press conference. Grazie onorevole. Ευχαριστώ κυρία Χάρμς. Αν είστε έτοιμοι θα ξεκινήσουμε τις ψηφορίες. Relazione McIntyre. Έκθεση McIntyre. Θα περιμένω ακόμα για λίγο μέχρι να καθίσουν όλοι οι συνάδελφοι και να προετοιμάσουν την κάρτα για την ψηφοφορία. Πρώτη έκθεση λοιπόν Μακιντάρ, έκθεση Μακιντάρ, πρόγραμμα ανταλλαγών, συνδρομής και κατάρτισης για την προστασία του ευρώ από την χαρα... παραχάραξη και την κυβδηλία. Πρόγραμμα Περικλής. Ονομαστική ψηφορία, έναρξη ψηφορίας, πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Έκθεση Ζάλμπα. Ζάλμπα. Ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Έκθεση Τζούμπερ. Ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Έκθεση πορέμπα. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Έκθεση νήτρας, ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Έκθεση Χιούμπνερ. Ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Επόμενη έκθεση. Έκθεση Μίτσελ. Ο εισηγητής παρακαλώ. Il relatore vuole parlare. Ο συγητής θέλει να μιλήσει. Κύριε Μίτσελ, απουσιάζει. Ε, ωραία. Τότε θα ψηφίσουμε. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Έκθεση Αγιάλα. Ορισμός μέλους του ελεκτικού συνεδρίου Φιλουίν Όεν. Μυστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται ο ορισμός. Ο ορισμός μέλος του ελεκτικού συνεδρίου, πάντοτε Αγιάλα, Άλεξ Μπρένικ Μέγερ. Μυστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Άλλος ένας ορισμός μέλους ελεκτικού συνεδρίου Έκθεση Αγιάλα. Ανδρή Γκρετέν. Μυστική ψηφοφορία. Άρχεται. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Άλλος ένας διορισμός μέλους του Ελευθερικού Συνεδρίου, ο κ. Νικόλας Μιλιώνης. Μυστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται άλλος ένας ορισμός, Ντανιέλ Λεμάρκ, μυστική ψηφοφορία, άρχεται. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τώρα έχουμε τον ορισμό του Προέδρου του Εποπτικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζα. Έκθεση Μπόζ, Ντανιέλ Νουή. Μυστική πάντοτε ψηφοφορία. Είναι μια γυναίκα, δώσαμε μεγάλη μάχη, παρόλο που δεν βρίσκεται στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, άρχεται η ψηφοφορία, πέρας της ψηφοφορίας, εγκρίνεται. Relazione Brock. Έκθεση Brock. Τροπολογία 1. Ποιο είναι υπέρ. Κατά. αποχέ εγκρίνεται. Πρόταση τη επιτροπή. Ποιο είναι υπέρ. Κατά. αποχέ εγκρίνεται. Νομοθετικό ψήφισμα. Ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα τη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Έκθεση Beauty Coffer. Τροπολογία 1. Ποιο είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Πρόταση της Επιτροπής υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Νομοθετικό ψήφισμα, ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Έκθεση Κούκαν, τροπολογία 1. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Πρόταση της Επιτροπής υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Νομοθετικό ψήφισμα, ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνεται έκθεση Ρούτσεκ, τροπολογία 1, ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται, πρόταση της Επιτροπής υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται, ονομαστική ψηφοφορία για νομοθετική πρόταση, άρχεται, πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνεται. Έκθεση Λόπες Ιστούριθ. Τροπολογία 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Πρόταση τη επιτροπή, Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Νομοθετικό ψήφισμα. Ονομαστική ψηφορία. Άρχεται ψηφορία. Πέρας εγκρίνεται. Έκθεση Λάμστορφ. Τροπολογία 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Πρόταση Επιτροπής. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται νομοθετικό ψήφισμα ονομαστική ψηφορία άρχεται η ψηφορία πέρας της ψηφορίας εγκρίνεται έκθεση Μπέρμα τροπολογία 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται πρόταση της Επιτροπής υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται νομοθετικό ψήφισμα ονομαστική ψηφοφορία άρχεται η ψηφοφορία πέρας Εγκρίνεται. Το λόγο έχει η Επιτροπή. Η Επίτροπος Βασιλείου. Κύριε Βασιλείου, έχετε το λόγο. Honorable members, Αξιότιμα μέλη, η Κομισιόν χαιρετίζει την έγκριση του Κοινοβουλίου για το μηχανισμό χρηματοδότησης ε, της υπηρεσία υπηρεσίας εξωτερικής που θα δώσει τη δυνατότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση να συνεχίσει να είναι παγκόσμιος παίκτη προάγοντας ε, τα συμφέροντα και τις αξίες του. Η δημοκρατία, η ειρήνη, η αλληλεγγύη, η σταθερότητα και η μείωση της φτώχειας όπως και η διασφάλιση παγκόσμιων ε, κοινών αγαθών θα είναι στην καρδιά της εξωτερικής δράσης την επόμενη επταετία. Τα μέσα μας δίνουν τη δυνατότητα να ε, συνεργαζόμεθα με τους εξωτερικούς εταίρους σε τέσσερις προτεραιότητες. Διεύρυνση, γειτονία, συνεργασία και στρατηγική εταίρη και ανάπτυξη της συνεργασίας. Εξ ονόματος Ευρωπαϊκής Επιτροπής επιθυμώ να ευχαριστήσω όλους τους εισηγητέ, όπως και εκείνου, που ήταν οι προκάτοχοί του για την επικοδομητική συμβολή του στι διαπραγματεύσει. Θα πρέπει να είμαστε περήφανοι για αυτό που επιτύχαμε από κοινού. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ κυρία Επίτροπε. Έκθεση Χάρκιν. Πρώτο τμήμα. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Πρόταση της Επιτροπής. Υπέρ. Κατά. Όχι. Συγγνώμη λέει πρόεδρος. Ωραία. Λοιπόν, πρόταση της Επιτροπής εγκρίνεται. Νομοθετικό ψήφισμα, ονομαστική ψηφοφορία, άρχεται, πέρας. Εγκρίνεται. Εκθεση Πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 8. Υπέρ κατά αποχές θα πρέπει να ελέγξουμε ηλεκτρονικά για την τροπολογία 8. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 12. Ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 14. Τροπολογία 14. Ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. 17. Πρώτο τμήμα. Ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, ονομαστική ψηφορία, άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 20, ονομαστική ψηφοφορία, άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 22, ονομαστική ψηφοφορία, άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 28. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Έλεγχος. Σηκώστε μου σας παρακαλώ τα χέρια. Άρχεται η ψηφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 29. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 30 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 31 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 26 ονομαστική ψηφοφορία άρχεται. Πέρας απορρίπτεται. 27 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται πρόταση της Επιτροπής. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Νομοθετικό ψήφισμα. Ονομαστική ψηφοφορία άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Ο εισηγητής επιθυμεί το λόγο. Πολύ σύντομα κυρία Πρόεδρε, εξηγώ ότι η ομάδα μου αποφάσισε να απόσχει στην τελική ψηφοφορία γιατί πιστεύουμε ότι είναι δίκαιο να δώσουμε πράσινο φως στην Επιτροπή για διαπραγματεύσει με το Συμβούλιο. Παρόλα αυτά είναι λυπηρό ότι το ΕΛΚ αποφάσισε να αποδυναμώσει την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που σχεδιάστηκε και υποβλήθηκε μετά από αίτημα της πλειοψηφίας των κρατών μελών το Μάιο. Ευχαριστώ. Ωραία. Έκθεση Κόβαξ. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 51. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 52. Ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 53. Ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 54. Ονομαστική. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 55. Ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. 37. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 56. Καταπίπτει 56. 57. Ονομαστική. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. 61-63 μέχρι 65 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται 58-60 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται 45 καταπίπτει και οι επόμενες πρόταση της Επιτροπής ποιος είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται νομοθετικό ψήφισμα, νομαστική ψηφορία άρχεται πέρας Εγκρίνεται. Έκθεση Κούκαν. Τροπολογία 7. Υπέρ. Σηκώστε τα χέρια σας παρακαλώ. Κανείς δεν είναι υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 8. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 9. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Παράγραφος 10 του αρχικού κειμένου σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, θα πρέπει να λέξουμε ηλεκτρονικά. Για το δεύτερο τμήμα άρχεται η ψηφοφορία, πέρας, εγκρίνεται. Δέκα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Ε, συγγνώμη, απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα, υπέρ. Καταπίπτωνο, καταπίπτωνο, συγγνώμη λέει η πρόεδρος, καταπίπτωνο τα υπόλοιπα τμήματα. 11, πρώτο τμήμα, υπέρ. Κατά, αποχές, απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα, υπέρ. Κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 2, υπέρ. Κατά, αποχές, απορρίπτεται. Έλεγχος ηλεκτρονικός για την τροπολογία 2. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Εγκρίνεται. 19. Τροπολογία 19. Σας παρακαλώ πολύ να τα χέρια. 19. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 12. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 27. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 30. Υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 13, πρώτο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές, ηλεκτρονικός έλεγχος, άρχεται η ψηφοφορία, πέρας, απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 15, πρώτο τμήμα, υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τρίτο Δέκα 16. Να λέξουμε ηλεκτρονικά, αλλά για ποιο τμήμα θέλετε. Για το δεύτερο τμήμα. Ωραία. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 16. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 43. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Να ελέξουμε. Για το δεύτερο τμήμα. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 6. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Α, με συγχωρείτε λέει πρόεδρος. Μόνο, μόνο η 6. Μόνο η τροπολογία 6. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 47 για το πρώτο τμήμα. Ποιο είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 14. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται 17 πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τρίτο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 18 θέλετε να λέξουμε για το τρίτο τμήμα ωραία, ωραία θα λέξουμε ηλεκτρονικά άρχεται πέρας όπως λέγαμε απορρίπτεται 18, τροπολογία 18 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 55, ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, να ελέξουμε. Άρχεται η ψηφοφορία, πέρας της ψηφοφορίας, εγκρίνεται. Τροπολογία 23. Έχουμε μια προφορική τροπολογία του εισηγητή. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Η τροπολογία που παρουσίασα είναι η εξής. Υπενθυμίζει τα ψηφίσματα της 25ης Νοεμβρίου 2010 για την κατάσταση στη Δυτική Σαχάρα, της 22ης Οκτωβρίου 2013 για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην περιοχή του Σαχέλ ε, ζητεί την εξασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για τους Σαχράουι και η ανάγκη ε, να καλυφθούν τα δικαιώματα αυτά στην Δυτική Σαχάρα και η ελευθερία ε, του συνέρχεστε και το δικαίωμα διαδηλώσεων και ζητάει την απελευθέρωση όλων των Σαχράουι πολιτικών κρατουμένων. Ζητάει το άνοιγμα του εδάφου σε ανεξάρτητους παρατηρητές μη και στα μέσα. Υποστηρίζει μια λύση πολιτική αποδεκτή από όλους για την Δυτική Σαχάρα σύμφωνα με τις, τα αντίστοιχα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών ακόμη και αυτών που επιτρέπουν την αυτοδιάθεση. Αυτή είναι η τροπολογία και ζητώ να την υποστηρίξετε. Ευχαριστώ. No. Quindi chi è a favore, chi è contro, chi si astiene, approvato. Per κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 3. Έχουμε μία προφορική τροπολογία κοπά. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα θέλαμε εξ ονόματος ε, της Σοσιαλιστικής και Δημοκρατικής Ομάδας να έχουμε μια τροπολογία. Καταδικάζει ε, την ε, στρατιωτική χρήση και τις ε, σφαγές με στόχο ως βασική παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ζητά να σταματήσουν αυτές οι δραστηριότητες και να έχουμε μια κοινή θέση σχετικά με τα drones, με τα μη επανδρομένα αεροσκάφη. Υπάρχουν αντιρρήσεις για αυτή την προφορική τροπολογία. Αν υπάρχουν θα πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον 40 ευρωβουλευτές που θα αντιτίθενται. Έτσι. Ψηφίσουμε το αρχικό κείμενο Τη τροπολογίας 3. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ωραία, αλλά έχουμε ηλεκτρονικά. Τροπολογία 3. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τώρα θα ψηφίσουμε το αρχικό κείμενο. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Θα πρέπει να ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Δεν είναι σαφές το αποτέλεσμα. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Ε, εμενταμέντο 20. Chi a favore? 20. Ποιος είναι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 4 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Αρχικό κείμενο παράγραφος 67 ποιος είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 5 ποιος είναι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 21. Να ελέξουμε το 5. Ωραία. Άρχεται η ψηφοφορία για την 5. πέρα της ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Ζητώ συγγνώμη, λέει η Πρόεδρος. Τροπολογία 21. Ποιος είναι υπέρ. Κατά απόχέ. Ελεκτρονικά θα ψηφίσουμε, δεν είναι σαφέ το αποτέλεσμα. Τροπολογία 21. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. Εγκρίνεται. Τροπολογία 22. ποιο είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 88 το αρχικού κειμένου υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 100 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 103 πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 116 πρώτο τμήμα ονομαστική ψηφοφορία, άρχεται η ψηφοφορία, πέρας, Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 119. Ονομαστική ψηφοφορία. Όχι, διορθώνει τώρα η πρόεδρος. Ένα λεπτάκι, να το κοιτάξω καλά, λέει η πρόεδρος. 118. 118 λέει τώρα. Ονομαστική ψηφοφορία. Πρώτο τμήμα. Ενάξι, Πέρας. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 119 ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 1. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Κύριε Κάσμα θέλετε το λόγο Ναι παρακαλώ Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε Κυρία Πρόεδρε ζήτησα να ελέγξω με την τροπολογία 20 το φώναξα δεν ακούσατε πιστεύω ότι υπήρχε πλειοψηφία υπέρ μπορούμε να επανελέγξουμε την τροπολογία 20 λοιπόν. Ευχαριστώ. Πολύ ωραία. Θα ελέξουμε την τροπολογία 20. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία για την τροπολογία 20. Τη βρήκατε την 20, ρωτάει πρόεδρος, πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Πολύ ωραία. Τελική ψηφορία υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Παρακαλώ. Κυρία Πρόεδρε, με συγχωρείτε για τη διακοπή ως σκιώδης για την ομάδα μου. Θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον συνάδελφο Τρεμόζα για την εξαιρετική συνεργασία για την ετήσια έκθεση. Δυστυχώ στον κατάλογο ψηφοφορία τη ομάδα μου υπάρχει ένα μικρό λάθο. Όταν ψηφίσουμε στην παράγραφο 73 και την τροπολογία 5, η ομάδα του Λαϊκού Κόμματος θέλει να προσθέσει αποχή. Έχει ε, σημειωθεί λάθος εκεί. Πολύ ωραία. Ευχαριστώ. 11. Αρχικό κείμενο. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 18. Ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 2 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 3. Έλεγχος. Έλεγχος για το 2. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Είχατε δίκιο. Απορρίπτεται. Τροπολογία 3. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Θέλετε λέ, να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Ωραία. 3 για την 3. Άρχεται. Πέρας. Αυτή η φορά είχα δίκιο εγώ λέει η Πρόεδρος. Ωραία. 30. Πρώτο τμήμα. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα ονομαστική ψηφοφορία. άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται 31. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 36. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 47 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 51. Θέλετε έλεγχο για την 47. Ωραία. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 51. Ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. 52 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 55. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 63. Τσέκ για το δεύτερο τμήμα, έτσι. Ωραία. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Δεύτερο. 63. Πρώτο τμήμα, λέει ο Πρόεδρος. 63. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα τη 63. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 64. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά αποχές φαίνεται να απορρίπτεται. Αλλά αν θέλετε μπορούμε να ελέγξουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 4. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τσεκ για το 5. 5. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 1. Ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται 93 το πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 105. Υπέρ. Κατά αποχές θα ελέγξουμε. Άρχεται η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Πέρας απορρίπτεται 108 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται ονομαστική ψηφοφορία για την τελική ψηφοφορία για το σύνολο άρχεται πέρας εγκρίνεται Ντόρφμαν τροπολογία 1 ονομαστική ψηφοφορία άρχεται η ψηφοφορία πέρας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 <clears throat> Κυρία Πρόεδρε, δεν θέλω να σας καθυστερήσω, αλλά είναι πολύ σοβαρό το θέμα. Χθες ε, στην έκθεση Εστρέλα ε, γράφτηκα ότι ψήφισα υπέρ της τροπολογίας του ΕΛΚ, ενώ εγώ ψήφισα κατά. Υπέπεσε στην προσοχή μου ότι ένα μέλος είχε παρόμοια εμπειρία. Γι' αυτό ζητώ από τις υπηρεσίες να κάνουν μία πλήρη έρευνα για να βεβαιωθούμε ότι το σύστημα ε, ψηφοφοριών ε, αντικατοπτρίζει πιστά τις ε, ψήφους της προτιμήσεις των μελών. Ευχαριστώ. Μου λένε ότι έχει ήδη γίνει και θα πρέπει να αποσταλούν οι ανακοινώσεις αυτές τις υπηρεσίες της αρμόδιες. Έκθεση Μίτσελ, 31 για το πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Θέλετε να αλλάξουμε τι, το 2, το 2 θέλετε να αλλάξουμε, ωραία, το ελέγχουμε. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Ehm, Ωραία, έκθεση Βερτμάν. Η εισηγήτρια έχει το λόγο. Non Απουσιάζει, εδώ δεν είναι, ναι. κυρία Βέρτμαν. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Πρόκειται για γυναίκες με αναπηρία. Καταλαβαίνετε πόσες ε, πολλαπλές διακρίσεις υφίστανται. Είναι 18 εκατομμύρια ανάπηροι ε, και 80% ε, ανάπηροι, 76 γυναίκες. Είναι κρίμα που δεν είχαμε παρά μόνο μια σύντομη συζήτηση. Ελπίζω η ψήφος στην έκθεση αυτή να είναι θετική. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Λεκή Πρόεδρος. 24 πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα ονομαστική ψηφοφορία άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 25 πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 26 πρώτο τμήμα υπέρ κατά Αποχέ εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά απόχέ εγκρίνεται. 47 πρώτο τμήμα υπέρ κατά απόχέ εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά απόχέ εγκρίνεται. 52 πρώτο τμήμα υπέρ κατά απόχέ εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά Αποχέ εγκρίνεται να ελέξουμε το δεύτερο τμήμα της 52 άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Το H, πρώτο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίνεται. Το 2, υπέρ, αποχές. Εγκρίνεται. Τελική ψηφορία, υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίνεται. De Jong, 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 10 πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τρίτο ονομαστική ψηφοφορία άρχεται πέρας εγκρίνεται 14 Πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 15. Ποιος είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 16. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα ονομαστική ψηφοφορία άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Τέταρτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Γκέμπαρτ, θέλει το λόγο, παρακαλώ. Το μικροφωνό σας. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Προέκυψε λάθος στον κατάλογο ψηφοφοριών μας. Η ομάδα μας θέλει να ψηφίσει κατά του δεύτερου τμήματος του 26 αρνητικό πρόσημο παρακαλώ. Ωραία, ευχαριστώ. 26. Πρώτο τμήμα, υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, υπέρ. Κατά αποχές. Να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά για το δεύτερο τμήμα. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 35. Υπέρ κατά Αποχές εγκρίνεται. Τελική ψηφορία υπέρ κατά. Αποχές εγκρίνεται. Θέλετε να ελέγξουμε. Όχι έτσι. Σας ευχαριστώ όλους.